ανοίγει διόδους που μπορούν να βρουν απαντήσει όσον αφορά το πρόβλημα της φορολογίας και ελπίζω να υιοθετήσει αυτή την έκθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε τον κύριο Ιβο Στρέιτσεκ